Γεια σας, καλώς ήρθατε σε αυτή την κοινή συνεδρίαση. Έκον Γιούρι. Θα συζητήσουμε πολύ σημαντικό ζήτημα για το Κοινοβούλιο που αφορά τις εκθέσεις αναχώρα εξετάζουμε τις 272 τροπολογίες που έχουν υποβληθεί σχετικά με αυτή την έκθεση. Θα ξεκινήσει η συζήτηση. Η Εύελιν Ρέγνερ και εγώ συμπροεδρεύουμε. Θα δώσουμε το λόγο στους συνεισηγητές που εκπροσωπούνται και δύο από την Εύελιν Ρέγνερ. Έχει πολλαπλές ιδιότητες σήμερα η Εύελιν. Έχει το λόγο Εύελιν. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε Ευχαριστώ και καλημέρα σε όλους και ξεκινάω κατευθείαν με, κατευθείαν τα γερμανικά γι' αυτό παρακαλώ να φορέσετε και τα ακουστικά σας εάν δεν ξέρετε γερμανικά. Ε, λαμβάνω λοιπόν το λόγο και ως εισηγήτρια και εκ μέρους ε, του Hugues Μπαγιέ με τον οποίο είχα μια πολύ καλή και στενή συνεργασία. Έτσι λοιπόν ε, αυτά που έχω να πω σε σχέση με τις μέχρι τώρα τροπολογίες εκφράζουν και τον κύριο Μπαγιέ και εμένα τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε καλύψει όπως είπε και ο Ρομπέρντο. 238 είναι οι τροπολογίες που έχουμε μέχρι τώρα κατατεθεί. Σημαντικός όγκος. Παρότι από πλευράς μας δεν υπήρξε μεγάλη, ε, μεγάλος αριθμός τροπολογιών, δεν είναι άλλωστε και η έκθεση μακροσκελής. Ε, τις τροπολογίες μπορώ να τις χωρίσω σε τέσσερις ομάδες εκείνες που μπορώ εύκολα να συνδυάσω ε, σε τομείς, δηλαδή, γιατί έχουν τα ίδια θέματα λίγο πολύ. Καταρχάς, το όριο 48β 40 αντί για 750 εκατομμύρια ευρώ ως όριο για την υποχρέωση. Τεράστια όμως η διαφορά, αν κοιτάξουμε τις, ε, τους ορισμούς και τα ποσά από την άλλη ευνόητη γιατί βλέπουμε δύο τάσεις. Αφενός με εκείνες τις τροπολογίες οι οποίες αναφέρονται στο νέο αυτό όριο των 750 εκατομμυρίων ευρώ για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία με την νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και βεβαίω φαντάζομαι θα λάβουν το λόγο οι συνάδελφοι για να εκθέσουν τι επιλογέ του. Αλλά βλέπω γενικά ότι είναι του ΕΛΚ, του ECR, οι τροπολογίε αυτέ. Με βάση την αρχή δηλαδή του BEPS, προσανατολίζονται στα 450 εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών, ενώ οι άλλες τροπολογίες, πάνω απ' όλα συναδέλφων από τους πράσινους, την ΚΟΕ, μέλη της ECR και από το FTD, αναφέρονται σε ένα κύκλο εργασιών ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ. Θα ήθελα αν προκειμένου να επισημάνω, και βεβαίως το βλέπουμε σε ορισμένες τροπολογίες, ότι στην οδηγία για τη λογοδοσία, για, τους, για τα λογιστικά accounting directive, αυτή η πρόταση της Επιτροπής θα επανέλθει με νομικό ορισμό. Θα ε, προβλέπεται λοιπόν ένας νομικός ορισμός του τι συνιστά μεγάλη, large, επιχείρηση και ποια είναι η μικρή. Είναι βέβαιο ότι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέχρι 40 εκατομμύρια ευρώ καθαρό κύκλο εργασιών αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Μέχρι εκεί οπωσδήποτε μπορώ να δώσω απάντηση για τις τροπολογίες που έχουν ε, κατατεθεί Απόλυτα είναι ξεκάθαρο ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής, δεν καλύπτονται από την οδηγία, μόνο οι μεγάλες. Άλλες τροπολογίες που κάνουν ε, παραπομπές σε θέματα χρηματοοικονομικά, ε, νομισματικά, ιδιαιτέρως ε, θα είναι χρήσιμες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για να επιτύχουμε συμφωνία και θέλω να ευχαριστήσω έτσι τους συναδέλφους που έχουν, τους που έχουν καταθέσει αυτές οι πληρωματικές ε, προ, ε, τροπολογίες οι οποίες μας ε, εμπλουτίζουν στην προσπάθειά μας και μας βοηθούν. Ένα δεύτερο μεγάλο μπλοκ τροπολογιών, ένα μεγάλο δηλαδή πολιτικό ζήτημα που αφορά την έκθεση και που βεβαίως καλύπτεται με τροπολογίες των συναδέλφων, είναι αυτό της πραγματικής έκθεσης φορολογικών στοιχείων αναχώρα που διακρίνεται από την έκθεση αναχώρα συν έκθεση φορολογικού παραδείσου. Δηλαδή γίνεται μια αντιπαραβολή σε σχέση με αυτό που είχε προτείνει η Επιτροπή στην έκθεσή της. Η υποχρέωση λοιπόν έκθεσης που προτείνει η Επιτροπή έχει να κάνει με τις δραστηριότητες και τις θηγατρικέ της επιχείρηση μέσα σε ένα κράτος μέλος συν ε, του φορολογικού παραδείσου. Αυτή είναι η μία ομάδα τροπολογιών που έχουμε λάβει, αλλά από την άλλη υπάρχει και άλλη μια μεγάλη ομάδα τροπολογιών που αναφέρεται σε στόχο μιας γνήσιας αναφοράς ή έκθεσης, δηλαδή έσοδα και φόροι από κάθε κράτος το οποίο έχει θυγατρική ή υποκατάστημα μια επιχείρηση. Και εδώ θα ήθελα να επισημάνω, ότι θα είναι άλλωστε σε όλους γνωστό, ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ήδη από την Επιτροπή Ανάπτυξης με την ψηφοφορία της προηγούμενης εβδομάδας σε θέματα που έχουν βεβαίω αναπτυξιακό καθαρά χαρακτήρα ή επιτοπλίστων χαρακτήρα. Και εκεί βλέπω ότι τα δεδομένα των ε, επιχειρήσεων υποστηρίζεται να αναφέρονται για όλες τις, επιχειρή... για όλες τις χώρες. Άρα λοιπόν μπορούμε να δούμε και αυτή την αναπτυξιακή περισσότερο προσέγγιση, έκθεση για όλες τις χώρες. Τρίτος τομέας, ξέρω ότι έχω ξεπεράσει τα πέντε μου λεπτά, αλλά μια και δεν είναι εδώ ο ΙΓ, λίγο πολύ θα καλύψω και το δικό του χρόνο. Όπως είπα και μαζί εργαστήκαμε και μαζί διατυπώσαμε θέσεις ε, και προτάσεις. Επιτρέψτε μου λοιπόν να αξιοποιήσω το δικό του μερίδιο του χρόνου. Τρίτος και μεγάλος τομέα, το περιεχόμενο, το περιεχόμενο των εκθέσεων κατά ανακράτος, τι στοιχεία θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και βεβαίως αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο αφετηρίας που γνωρίζουμε από την BEPS. Ε ε, διαφορετικά στοιχεία, ε, πολλά είναι αναλυτικά στοιχεία που μας ζητούν ορισμένες τροπολογίες, μπορούν να αλλάξουν δηλαδή τελείως την προσέγγιση και με ενδιαφέρει να δω και πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Όπως είπα, είναι πολλές προτάσεις που ζητούν περισσότερο περιεχόμενο, πιο πλούσιο περιεχόμενο, ενώ κάποιες άλλες τροπολογίες που ζητούν συγκεκριμένα και λίγα στοιχεία. Περιμένω λοιπόν να ακούσω τι έχετε να μας προτείνετε και εσείς με πολύ ενδιαφέρον. Φυσικά απαραίτητα είναι τα στοιχεία της επωνυμίας, της γεωγραφικής έδρας, η έκτασης, ε, πωλήσει, αλλά και άλλα όπως πωλήσει, αγορές, ενεργητικό, κόστος λειτουργίας. Όλα αυτά ίσως μπορούμε να τα δούμε με τη συζήτηση στη συνέχεια. Ποια σημεία δηλαδή θεωρείται πολύ σημαντικά και ποια θα μπορούσαμε ίσως να αφήσουμε κατά μέρος. Τέταρτος τομέας, τέταρτο η ομάδα, ε, Open Data Format, δηλαδή ο μορφότυπος ενιαίου εγγράφου, ένα μητρό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή με βάση το οποίο θα καταγραφόνται τα στοιχεία. Εδώ έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες τροπολογίες. Λάβει. Δηλαδή, και πάλι μπορούμε να βρούμε κάποιες λύσεις συνεργασία με τους συναδέλφους. Ε, τώρα για να συνοψίσω, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι Βλέπουμε από τις ε, τροπολογίες πως ε, υπάρχουν ε, τοποθετήσεις που ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση από τη μία ή την άλλη πολιτική ομάδα, ενώ άλλες οι οποίες είναι μεταξύ τους αντιφατικές. Και βέβαια καθήκον μας ως εισηγητών, αλλά και σκιωδών εισηγητών, είναι να συγκεράσουμε συνδυάζοντας και ανταλλάσσοντας θέσεις από τον ένα ή τον άλλο τομέα. Γι' αυτό λοιπόν θέλω σήμερα να δούμε τι προτείνουν, ε, τι θεωρείται ως απολύτως απαραίτητο, γιατί οπωσδήποτε θέλουμε μια γνήσια δημόσια, δημοσιοποίηση συγγνώμη, ε, ανά χώρα Θέλουμε μια δουλειά που θα γίνει καλά από το Κοινοβούλιο, που θα είναι χρήσιμη και που θα μπορέσει να μας βοηθήσει και στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, γιατί ξέρουμε το Συμβούλιο για ορισμένα ζητήματα μάλλον τραβάει το φρένο. Και γι' αυτό θα ήθελα με πολύ ενδιαφέρον να ακούσω τις δικές σας προτάσεις και παρατηρήσεις, ελπίζοντας πως εν τέλει, εν τέλει το Συμβούλιο θα αντιμετωπίσει μια θέση δική μας, ε, ισχυρή και ενωμένη. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε τώρα. Ο κ. Ροζάτη είναι ο πρώτος ομιλητής για τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, και προς τους συνεισηγητές. Αλλά ευχαριστούμε για τη συνεργασία και τους σκιώδες συζητητές έδειξε η Κομισιόν ότι έχει πάρει στα σοβαρά το θέμα της βελτίωσης των φορολογικών συστημάτων και να περιοριστεί η φοροδιαφυγή, οι απάτες και βέβαια και το ΕΛΚ είναι αναφανδόν υπέρ. Όμως, ο φάκελος αυτός τον οποίο σήμερα συζητούμε θεσπίζει την δημοσιότητα και δημοσιοποίηση των φορολογικών δεδομένων για να έχουμε περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τις ε, φορολογικές υποχρεώσεις των εταιριών στην Ευρώπη. Θέλουμε ότι αυτός ο στόχος είναι θεμητός, αλλά θα μην εξισορροπηθεί με έναν άλλο σημαντικό στόχο που είναι το να παραμείνουν οι εταιρείε μας ανταγωνιστικές. να μην προσθέτουμε επαχθείς διαδικασίες όπως αυτές τις κοινοποιήσεις. Υπάρχει βέβαια μπροστά μας η πρόκληση να βρεθεί αυτή η ισορροπία μεταξύ του ότι χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια από τη μία και από την άλλη μεριά η προστασία των εταιριών μας. Να μην τις στριμώχνουμε και έτσι να έχουν μειονέκτημα σε σχέση με τους μη Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους. Πιο συγκεκριμένο τώρα. Συμφωνώ 100% με την προλαλή σας ότι έχουμε 4-5 σημεία όπου ακόμη δεν έχουμε συμφωνήσει. Να σας πω τι πρεσβεύει το έλεγχο σχετικά. Πρώτα αυτό το 750 BEPS ως κατόφλι για αναπτυγμένε χώρε και για αναπτυγμένε ε, χώρε και ευρωπαϊκέ χώρε σε σχέση με, με τα 4 εκατομμύρια. Ε, ε, εντάξει, εμεί με το 750 και τίποτα δεν θέλουμε να παραβλάψουμε το πρότυπο το οποίο συμφωνήθηκε μετά από τι διαπραγματεύσει των ΩΣΑ. Από τα Μακρέ, επίση δεν θέλουμε να έχουμε επιπλέον βάρη για τι ευρωπαϊκές εταιρείε που θα τις κάνουν να στερούν τον Επίση, το ποιο θα είναι το εύρος, το, μέχρι πού θα φτάνουν αυτές οι πληροφορίε να περιοριστούν αυτά τα οποία απαιτούνται από τις εταιρείε και οπότε θέλουμε να υπάρχει ένας περιορισμός η αυστηρά στα όσα ε, το Action 13 του BEPS ε επιτάσσει. Επίσης ε, αυτού του είδους ο διαχωρισμός για τις εκθέσεις έχουμε μόνο τις εταιρείε που είναι σε list δηλαδή αυτές που είναι σε ε, φορολογούς παραδείδους, όχι άλλοι. Και επίσης να έχουμε αυτές τις ε, ρήτρες εξαίρεσεις για τις θηγατρικές. Η λύση εδώ δεν είναι εύκολη. Οι θηγατρικές εταιριών που είναι εγκατεστημένε σε άλλες χώρες, ΙΠΑ, Κίνα ή Καναδά, ίσως δεν θα μπορέσουν να παράσχουν τις πληροφορίες που πρέπει και αν δεν μπορέσουν να παράσχουν αυτά τα στοιχεία ε, τότε θα πλεονεκτούν έναντι των δικών μας εταιριών. και δύσκολα αυτό να συμφιλειωθεί με αυτό το οποίο θέλουμε να νομοθετήσουμε. Άρα αυτό δεν θέλω να σας επισημάνω. Είναι πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε. Και δεν έχει κριθεί οριστικά από μας το τι θα ψηφίσουμε πολλά βέβαια, θα εξαρτηθούν από τους συμβιβασμούς που ελπίζουμε να κλείσουμε με τους άλλους συνεισηγητέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ ο κύριο Γκουαλτιέρη. Ή, συ, όχι, όχι, όχι. Όχι, ο κύριο Γκουαλτιέρη διορθώνει. Πάμε πάλι στην Επιτροπή Νομική. Πού είναι, πότε θα έρθει η κυρία, αργότερα. Τότε, όντως, ECR λέρνερ Ευχαριστώ, πρόεδρε. Για αυτού του είδους την έκθεση αναχώρα, το επιχείρημα συνήθως ότι έτσι διαραίουν εταιρικά μυστικά. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό πλέον. Και μπορεί η ίδια η εταιρεία να δει τα οικονομικά στοιχεία και τα στατιστικά στοιχεία των ε, κυρίως εταιριών από άλλες χώρες. Αλλά τα ξέρουν αυτά και οι ανταγωνιστέ και αυτό το οποίο λείπει είναι η πληροφορία από αναπτυσσόμενες χώρες και από φορολογικούς παραδείσους. Άρα το εμπορικό απόρριτο δεν ισχύει για όλους. Έτσι να μπορέσουμε να φροντίσουμε την ανταγωνιστικότητα των εταιριών μας, άρα όλοι να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις για δημοσιοποίηση πληροφοριών και να ισχύει το, το, το ποσό των 40 εκατομμύριων που ήδη ισχύει. Να μην έχουν πλονίγμα οι μεγάλες εταιρείε τώρα. Το επιχείρημα των επιπλέον δαπανών για την κοινοποίηση των στοιχείων δεν ισχύει. Χρειάζονται στοιχεία αναχώρα. Και αυτό χρειάζεται για λόγους και λογιστικής και προγραμματισμού. Επίσης, ε, κατόφλη σε σχέση με το τζίρο όσον αφορά το διοικητικό άχθος. Πολλές εταιρείε ήδη συλλέγουν δεδομένα, απλώς δεν υποχρεούνται να τα κοινοποιήσουν. Άρα, το ότι υπάρχει διοικητικό άχθος δεν ισχύει. Και αυτή η κοινοποίηση αναχώρα έχει ζητηθεί και από άλλους εμπλεκομένους πέραν των ε, χωρών και θεσμικών οργάνων. Πολλοί επενδυτέ. Γιατί τον υπάρχουν αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ βασικά για τον κόσμο σε σχέση με τις εταιρείε. Και να είναι αυτά τα στοιχεία όσο γίνεται πιο ποιοτικά, όσο γίνεται. επίσης Επίση, χρειάζεται να υπάρχει αυτή η κοινοποίηση αυτών των στοιχείων, έτσι υπάρχει διαφάνεια, λειτουργεί καλύτερα η αγορά και ο ανταγωνισμός. Εμείς θέλουμε στο ECR καλύτερη λειτουργία της αγοράς, αλλά δεν συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι στην ομάδα με τις δικές μου απόψεις. Θεωρώ ότι αν ε, μόνο 10% της μεγάλης εταιρείας ισχύει αυτό το κατόφλι αυτό, έρχεται σε αντίθεση με τον ορισμό που δίνουμε στη μεγάλη εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, κάποιες εταιρείε τώρα θα έχουν συμπληρωτικό μειονέκτημα. Thank Σας ευχαριστώ. Δεν είναι εδώ και ο Σκαρίμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως και την τελευταία φορά θα μιλήσω και για τον κύριο Καβαντά. Δεν μπόρεσε να έρθει γιατί είναι στην καυτή προεκλογική εκστρατεία στη χώρα του. Άρα θα σας μιλήσω για λογαριασμό και των δυο μας, σαν τοποθέτηση των φιλελευθέρων. Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία για μας είναι το να γίνει κάτι, το να υπάρξει το υποσυζήτηση, το να υπάρξει μια τέτοια χειρονομία προς τον κόσμο, προς την κοινωνία και έτσι να πάμε προς περισσότερη διαφάνεια και να υπάρξουν οι απαραίτητες γνώσεις για δημοκρατική συμμετοχή. Βεβαίω και έχει αυτή η κίνηση πάρα πολλούς ε, εχθρούς κάποιες εταιρείε, προβλήματα στο Συμβούλιο, πάρα αυτά. Το έχω πει επανειλημμένα. Το καλύτερο είναι εχθρό του καλού. Άρα θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο και να μην ματιωθεί αυτή η πρωτοβουλία γιατί θα είναι πάρα πολύ κακό πολιτικά και αυτό θεωρούμε ότι είναι μια πρώτη διαδρομή, ένα πρώτο διεύμα και ότι υπάρχει κατάλληλη αναλογικότητα για να περάσει αυτό το οποίο έχει μπλοκαριστεί και να προχωρήσουμε. Οπότε έχουμε τώρα αυτούς τέσσερις βασικούς άξονες θέματα Οπότε θα πρέπει εδώ να, να τα βρούμε. Πρώτα πρώτα αυτό το κατόφλι, όπω είπε η συγκεκριτή. Εδώ δεν έχουμε τοποθετηθεί, φίλε Ελεύθερη. Έχουμε πει όμως το εξής και το επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για θέμα σχεδόν τεχνικό. Δεν έχουμε όλα τα στοιχεία. Παρακαλώ την Επιτροπή, παρακαλώ τους συνεισηγητές να τοποθετηθούν υπέρ των 40 εκατομμυρίων. Και δεν έχουμε τα στοιχεία για να μπορέσουμε να βρούμε ένα σημείο συμφωνίας, ένα σημείο ισορροπίας. Το θέμα είναι, που θέλουν πληροφορίε είναι το πόσο θα εκόστιζε. οι επιχειρήσεις σε σχέση με το 750. Να, ή αν κατέβουμε από το 750 στο 700. Από το 90 θα πάμε στο 97%. Ε, αυτό θα ήταν ενδιαφέρον, το ξέραμε. Και δεύτερον, ο μόνος κίνδυνος που διατρέχουμε, νομίζω, είναι ότι κάποια από τις μεγάλες γνωστές επιχειρήσεις που είναι στον τομέα των ΜΜΕ να διαφύγει να διαφύγει με το κατόφλι των 750. Πολυεθνική, ξέρω εγώ τι. Να την κλιτώσει με το 750. Άρα αυτό θα ήταν πάρα πολύ άσχημο σε σχέση με αυτό το οποίο επιζητούμε, δηλαδή να δώσουμε κάτι διάφανο στην ε, κοινή γνώμη. Δεν είναι το θέμα φορολογικό. Είναι θέμα διαφάνειας. Άρα η τάση μας είναι να συμφωνήσουμε με τον ΟΣΑ. Δηλαδή ε, ο ορισμός της μεγάλης εταιρείας όσον αφορά τις επιδοτήσεις, ενισχύσεις, ε, τώρα ε, είναι το μέγεθος το οποίο χρειάζεται να, να επικαλεστούμε εδώ όσον αφορά τη φορολογική αυτή Επίσης, ε, να μην ανοιχτεί η πόρτα όσον αφορά το να τα βρούμε τελικά, να τα βρούμε με βάση την λογική και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε. Δεύτερον, τι θα ε, πούμε και τι δεν θα πούμε. Δηλαδή τι θα ε, κοινοποιηθεί και τι δεν θα κοινοποιηθεί. Ε, όχι, κανένα ε, δεδομένο καινούργιο. Μα ήδη αυτά τα δίνουν στις φορολογικέ αρχέ. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Δεν θα γίνουν τίποτα καινούργια. Τώρα είναι μέσω αυτών των στοιχείων. Επίσης θα πρέπει με εξυπνάδα να φροντίσουμε να μην συρρυκνώσουμε την στρατηγική ικανότητα, την ικανότητα προγραμματισμού διείσδυση στην αγορά των εταιριών σε σχέση με τις άλλες. για να μπορέσει να λειτουργήσει εύρεθμα μια αγορά υπάρχει το βασικό κριτήριο, η αρχή της αμοιβαιότητα. που μην το κάνουμε μην ισχύει σχέση με Ιάπωνες, Αμερικάνους κλπ. Άρα εμείς μπορούμε να δώσουμε το πράσινο φω αν ισχύσει η λίστα του BEPS σε σχέση με το τι πρέπει να κοινοποιείται. Και να υπάρχει κάποια ρήτρα διαφύλαξη όσον αφορά σε σχέση με το μπορεί να ζητείτε να χρησιμοποιείτε μια υποπτική επιτροπή, να υπάρχει και να ζητηθεί ένας κατάλογος με αιτιολογήσεις, να δικαιολογήσει κάποιος δηλαδή κάποια στοιχεία αλλά να μην θεωρήσουν ότι παραβλάπτονται οι επιχειρήσει. Οπότε τότε θα προβούν σε περικοπές ή θα πάμε για να κατέβει το κατόφλι. Τρίτο Τρίτος και θέμα, η συγκέντρωση αυτών των στοιχείων. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε λογικοί, τα έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως με την έννοια του ότι γνωρίζει η Κομισιόν πόσο θα δυσκολευτεί πρόσθετο. Άρα, ίσως θα μπορούμε να έχουμε κάποιο άλλο σημείο συνάντησης και να αφήσουμε την πόρτα ανοιχτή, τη δυνατότητα δηλαδή ανοιχτή, να μπορέσει το Κοινοβούλιο, ή τέλο πάντων τα θεσμικά όργανα, να ζητούν πληροφορίες για, από κάποια συγκεκριμένη χώρα, κάποια συγκεκριμένη στιγμή, όταν δημιουργούνται υποψίες ή όταν αυτό θεωρείται λογικό να γίνει λόγω του κατάστασης κοινή γνώμης. Άρα θα πρέπει να δουλέψουμε με περισσότερη ευηλιξία. Και βέβαια θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της μαύρης λίστας. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ο Πρόεδρος. Και τώρα για την ΚΟΕ. Yes, you have the floor. Έχει το λόγο. Ναι κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς ο σκιώδης εισηγητής μας ο Μιγγέλ Βιάγας δεν μπόρεσε να έρθει. Εγώ θα τον αντικαταστήσω. Να σας διαβάσω τι πρεσβεύει για την έκθεση αυτή. Να τον συμπαθείτε. Τέλος πάντων, πρώτα-πρώτα, μπράβο στους συνεισηγητές. και αποφασίσαμε να μην κατεβάσουμε τροπολογία όσον αφορά τα κατόφλια και όσον αφορά την ε, κατάρτιση, την ανάλυση των ε, δεδομένων. Θα πρέπει όμως να σκεφτούμε ότι αυτά τα οποία λέει η Επιτροπή δεν αντεπούν τις προσδοκίες του κόσμου. Είμαστε υπέρ των 40 εκατομμυρίων. Και επίσης θα πρέπει να υπάρχει η κατάρτιση των κοινοποίησεων, των στοιχείων όπως είπαμε. Τώρα όσον αφορά τα κριτήρια διαβίβασης για να δούμε πώς θα πρέπει να αναδειχθεί το τι ισχύει τους εργαζόμενους ανά κλάδο. Η αρχική πρόταση των εισηγητών ήταν ε, εύστοχη, οπότε εμείς θα τα βρούμε, θα κατέληγουμε σε κάτι συμβιβαστικό. Συμφωνούμε επίσης ότι θα πρέπει να έχουμε κάποια κοινή πλατφόρμα αλλά θα πρέπει να δούμε πώς οι διάφορες φορολογικές αρχές θα συντονίζονται. Και αυτό μέσω φορέων, οργάνων διακυβερνητικών. Σας ευχαριστώ. Πασκάλ Ντουρά. Πασκάλ Ντουρά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να υπενθυμίσω στον εισηγητή ότι χάρηκα που διάβασα αυτή την έκθεση. Πολύ ποιοτική δουλειά που έγινε. Τη χαιρετίζω. Και όπως και ο προλαλής σας της Γκουε, να πω και εγώ, ότι μας ικανοποιεί εν γέννη η έκθεση. Μας ικανοποιεί απόλυτα. Παρ' όλα αυτά, να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις του κ. Καθεσαμπό. Τις είχε θέσει και την προηγούμενη φορά εφόσον ζητά πρέπει να δοθούν κάποιες ε, διευκρινήσεις που είναι απλούστατες να δοθούν. Το πρώτο ερώτημα που τίθεται το θέμα είναι του κατοφλίου. Γιατί να κρατήσουμε τα 40 εκατομμύρια και να μην έχουμε τα 700 εκατομμύρια και τι συνέπειες επιφέρει αυτό. Δεν θέλω να απαντήσω για τους ηγητές, αλλά για να πούσω το λόγο. Διότι τα 40 εκατομμύρια σαν όριο είναι αυτό του ορισμού της, ε, αρχ... της ε, λογιστικής οδηγίας για τις μεγάλες επιχειρήσεις οριζόμεθα επιφυσταμένου ορισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τις μεγάλες επιχειρήσεις εν συγκρίση με τις λιγότερο μεγάλες. Γιατί αυτό το κατόφλι και όχι άλλο, διότι παραμένουμε στα πλαίσια της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου και δεν φεγραμμιζόμεθα απαραίτητα με τις θέσεις κάποιου διεθνούς οργανισμού που δεν λέω ότι δεν αξίζουν τον κόπο, αλλά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τους Ευρωπαίους νομοθέτες αυτοί οι φορείς. Αυτά για τα 700 εκατομμύρια. Εν συγκρίση με τα 40. Το δεύτερο ερώτημα του κυρίου Καλβέ Σάμπον και ξέρει την απάντηση, αλλά δεν πειράζει. Ας κάνουμε ότι δεν γνωρίζει τη διαφορά. Το όριο των 40 εν συγκρίση με τα 700 μας κάνει να πάμε το 90% των επιχειρήσεων που δεν θα ε, τις αφορούσε το κείμενο στα 90% που τις αφορά το κείμενο. Εν γέννη ε, πάμε από το 10% στο 90%. Κύριε Καλβέ Σαμπον, ε, πιστεύω ότι γνωρίζετε την κατάσταση. Λοιπόν, το θέμα του ορίου αυτού είναι κάτι που δεν είναι αθώο και ανώδυνο. Θα πηγαίνω από το 10% στο 90% για να είμαστε αντικειμενικοί, απόλυτα αντικειμενικοί. Δεν είναι μόνο ο αριθμό των επιχειρήσεων ή των εταιριών που καλύπτονται που πρέπει να ληφθεί υπόψη, αλλά και ο τζίρο που αντιπροσωπεύει αυτό. Εκεί πράγματι θα καλύπταμε πάνω το 10% μέσω των 700 εκατομμυρίων, διότι μόνο οι πολύ μεγάλε επιχειρήσει έχουν το μεγαλύτερο τζίρο. Εν γέννη η συνέπεια είναι σημαντικότατη. Πρέπει να κατευθύνουμε προς ένα κατόφλιο που θα είναι εξελικτικό με την πάροδο του χρόνου, ε, εξελίξιμο, μπορούμε να το δούμε. Μπορούμε να βρούμε ενδιάμεσες λύσεις. Αυτά. Μακρο, μακρηγόρησα επ' αυτού, αλλά διότι προφανώς είναι σημαντικότατο. Μετά, το θέμα της συλλογής και σώρευσης των πληροφοριών. Το συζητήσαμε αυτό. Η συνεχής επικαιροποίηση του καταλόγου των φορολογικών παραδείσων είναι με δραστηριότητα σχεδόν αδύνατη, ενώ η διαφάνεια των πληροφοριών σε επίπεδο επιχειρήσεις αυτό είναι κάτι απλούστατο να εφαρμοστεί κατά χώρα. Έδωσε το παράδειγμα του Delaware στη ΣΥΠΑ. Πώς ε, να βάλουμε τη ΣΥΠΑ στις φορολογικούς παραδείσους. Αυτό δεν είναι λογικό, δεν είναι σοβαρό, ενώ το να ξέρουμε πόσα πληρώνει κανείς ε, φόρους σε μια πολιτεία των ΗΠΑ είναι κάτι απλούστατο για την επιχείρηση. Το διοικητικό άχθος, εκεί πρέπει να είμαστε σοβαροί, όσο έχουν τα πράγματα, οι συγμένες επιχειρήσεις που έχουν ε, στο διοικητικό του συμβούλιο ε, ανθρώπου του συστήματος πρέπει να, να αναφέρουν λεπτομερώς τα οικονομικά του στοιχεία. Η ομαδοποίηση των στοιχείων πολύ σημαντικό. Το πεδίο εφαρμογή το υποστηρίζω, χωρί επιστρέφω σε λεπτομέρειε. Το άλλο σημείο είναι πιο τεχνικό. Άκουσα τα διάφορα επιχειρήματα για τι πληροφορίε που να δίδονται. Ποιο είναι ο βαθμό των πληροφοριών που θα πρέπει να χορηγούνται και να εμφανίζονται στι λογιστικέ δηλώσει. Εκεί πρέπει να ομολογήσω αυτό το σημείο, χρειάζεται βάθυνση Όσο επισερχόμεθα στι λεπτομέρειε, τόσο η δουλειά των φορολογικών φορέων και των τρίτων θα διευκολύνεται. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πασκάλ. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο σε έναν εκπρόσωπο του EFTD. Η κυρία Φεράρα δεν είναι εδώ. Εσείς ποιος την εκπροσωπεί. Η Στόρχ, εγώ είμαι. Συστούμε σήμερα λοιπόν την άρση του φορολογικού απεωρήτου για τις επιχειρήσεις και έτσι έχω προς τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος το εξή ερώτημα. Τι πάθατε. Δύο συνεισηγητές ε, και οι δύο σοσιαλιστές συνήθως ε, προσπαθούν να ελέγχουν την κατάσταση οι συντονιστές και δεν καταλαβαίνω πώς σας ξέφυγε όλη αυτή η κατάσταση και έχετε ορίσει δύο εισηγητές ε, από τους σοσιαλιστές ή δεν καταλάβατε τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Είτε λοιπόν πρόκειται για ευρωπαϊκές, είτε πρόκειται για, από τρίτες, ε, για επιχειρήσεις από τρίτες χώρες, πρέπει αν έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 750 εκατομμύρια ευρώ να δημοσιεύουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Απίστευτο η Επιτροπή εδώ καταχράται των αρμοδιοτήτων της για τη δημοσιοποίηση προκειμένου να βάλει χέρι στην ε, φορολογική νομοθεσία η οποία είναι ουσιώδης ε, εθνική αρμοδιότητα και πρέπει να παραμείνει. Το μόνο λοιπόν το οποίο μπορώ να ε, συστήσω στις επιχειρήσεις είναι να προσφύγουν εναντίον της σχετικής νομοθεσίας όταν εγκριθεί για να την ακυρώσουν. Οι σοσιαλιστές βλέπουμε ότι θέλουν μια φορολογική αρμοδιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται ότι αδιαφορούν και για την παρανομία, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτό να συνεχιστεί. Πολλές φορές αναφέρθηκε επίσης ότι θέλετε να μειώσετε και το επίπεδο της υποχρέωσης ε, δήλωσης από τα 750 στα 40 εκατομμύρια ευρώ κύκλου εργασιών. Τι διαβάσατε την πρόταση της Επιτροπής. Γιατί την θεωρία αναλογική μόνο και μόνο επειδή ήταν πολύ υψηλό το όριο και επειδή αφορά μόνο μεγάλες επιχειρήσεις και όχι μικρές. Εκείνες δηλαδή τις οποίες ε, αφορά ούτως ή άλλως η οδηγία για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Δηλαδή εσείς μειώνετε αυτό το υψηλό ε, κατόφλι από τα 750 εκατομμύρια που έλεγε η Επιτροπή στα 40 και άρα πλήτεται τις μικρές επιχειρήσεις, πλήτεται την καρδιά της οικονομίας. Τι είναι αυτό, απλώς είστε κακοί, κακεντρεχείς έναντι της οικονομίας ή κρύβεται κάτι άλλο πίσω από αυτό. Ή αν είναι απλώς να παίξουμε την κολοκυθιά, να κάνω και εγώ τη δική μου συνεισφορά. Αντί να μειώσουμε από 750 εκατομμύρια στα 40 εκατομμύρια, ας αυξήσουμε από τα 750 εκατομμύρια στα 750 δισεκατομμύρια τον κύκλο εργασιών ω όριο. Και εν πάση περιπτώσει βλέπουμε εδώ πέρα πόσο παράλογο είναι αυτό. Όλοι αυτοί που προσπάθησαν να συζητήσουν βλέπουμε ότι έχουν παρετηθεί. Το Business Europe διαβάσατε τι μας έγραψε. Είναι εξαιρετική επιστολή για δύο λόγους. Καταρχάς διότι ξεκάθαρα λέει ότι βλέπει πως γίνεται συζήτηση και διαπραγματεύση κάτι το τελώς παράλογο. Μας το λέει ξεκάθαρα. Και δεύτερον, εξαιρετική είναι αυτή η επιστολή, διότι την παραγνωρίζετε. Διότι θα την αγνοήσετε, δεν θα την λάβετε καθόλου υπόψη και έτσι θα ξυπνήσουν και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι επικριτικές απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλες οι οποίες είναι θετικές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιληφθούν τι μεγάλο κακό κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό παρακαλώ τους συναδέλφους να υποστηρίξουν την πρότασή μου παριθμών 37, τροπολογία 37, για απόρριψη της πρότασης. Ευχαριστώ πολύ. Σκιώδης για το ΕΝΦ είναι η κυρία Κάπελ. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ η καταπολέμηση της φοροαποφυγής από το LuxLeaks και μετά είναι κύρια προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια στη φορολογική, στο φορολογικό ανταγωνισμό και την εφαρμογή των κανόνων της φορολογίας. Άρα η διαφάνεια έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε και την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και τις εκθέσεις στη δημοσιοποίηση φορολογικών στοιχείων ανακράτος. Ιδιαίτερα εδώ καλούνται οι αρχές των κρατών μελών να ενημερώνονται για τις δηλώσεις των επιχειρήσεων, κυρίως των μεγάλων επιχειρήσεων, των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ίσως λοιπόν θα ήταν καλό να τηρήσουμε τις αρχές του BEPS, του ΩΣΑ. Και άρα δεν υποστηρίζω την ιδέα της μείωσης του κατοφλίου των 750 εκατομμυρίων ευρώ σε 40 εκατομμύρια κύκλου εργασιών. Νομίζω ότι η δημοσιοποίηση ε, των φορολογικών στοιχείων είναι ήδη σοβαρή υπόθεση, έχουν την αρμοδιότητα, είναι στη διαθέση μάλλον των αρχών των κρατών μελών και σημαντικό είναι να δημοσιοποιείται, όπως ζητήσατε να σας πούμε, αυτό που προβλέπει ο κανόνας μπέπς στοιχεία τα οποία ούτως ή άλλων μπορούν διεθνώς να δημοσιοποιούνται για να διαφυλαχθεί και η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παράλληλο σεβασμό στην αρχή της διαφάνειας. Είναι σημαντικό να έχουμε διαφάνεια, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος ε, ε, του ανταγωνισμού και μάλιστα και του διοικητικού. Γι' αυτό λοιπόν ας είναι δημόσια τα στοιχεία, ας υπάρχει δυνατότητα της ανταλλαγής μεταξύ των δημοσίων αρχών των στοιχείων που είναι απαραίτητα, αλλά όχι στο δημόσιο. Μετά για τις αρχές, για τις τράπεζες, για τις φορολογικές αρχές, ναι μπορούν να διατίθεται τα στοιχεία, αλλά όχι στην κοινή γνώμη. Ευχαριστώ. Φεραγκούτ. Και μετά η κυρία Μπέρες. Ευχαριστώ πολύ. Όπω ξέρετε εμεί και ούτε για, για την νομική επιτροπή και η πρότασή μα και οι 22 μα τροπολογίες όπου προέρχονται από πολλού βουλευτέ. είμαστε υπέρ τη πρόταση τη ε, Κομισιόν για να βρεθεί μια ισορροπία όσον αφορά την διαφάνεια από τη μία αλλά και από την άλλη να υπάρχουν εγγυήσει ότι δεν θα παραβλαβεί το κλίμα το επενδυτικό στην Ευρώπη αλλά θα προστατεύσουμε και την ανταγωνιστικότητα για το φορμάτα να συμβαστούμε για την κοινοποίηση αναχώρα και να δούμε πώς θα βρεθεί συμβασμό μεταξύ των 750 και των 40. Υπάρχει εδώ πέρα μεγάλο περιθώριο. Και να λάβουμε υπόψη και τι προτείνει όσα στο Συμβούλιο. Μόνο η Ελλάδα έχει πει να μειωθεί το ποσό των 250 και κάποια άλλα που θέλουν απλώς να μπλοκαριστεί το νομοθέτημα. Αυτό το, να ξέρουμε όμως ε, πώς έχει συγκυρία και το περιβάλλον. Γιατί έχουν υπάρξει και άλλες νομοθετικές προτάσεις από διάφορες επιτροπές που τελικά μένουν στο ψυγείο. Ο κύριο Καλβέ ζήτησε περισσότερη ενημέρωση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και εγώ θα ζήταγα το ίδιο. Περισσότερα στοιχεία για να ξέρουμε ακριβώς σε τι περιβάλλον κινούμεθα. Περισσότερη διαφάνεια. Αυτό κάνει η Επιτροπή. Ακριβώ αυτό που ζητήσαμε και οι επιχειρήσει όμως ζήτησαν και γι' αυτό και κατεβάσαν και εμείς δύο τροπολογίε για μια ρήτρα διαφύλαξη Έτσι οι επιχειρήσεις όσον αφορά την κοινοποίηση των πληροφοριών όταν υπάρχει κίνδυνος ε, βλάβης της εμπορικής τους θέσης να εξαρτούν. Και αυτό είναι ε, κάτι πράγματα που τόσο ώστε να υπάρχει ισορροπή Και επίσης να δούμε θα γίνει τη διάρκεια της διαδικασίας ασφαλιαρική από μία, διαφάνεια την να δούμε το σωστή ισορροπή. Ευχαριστώ, Υπερβός. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πρότασή της. Υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι πρέπει να βρεθεί συμβιβαστική λύση μεταξύ 40 εκατομμυρίων και 750 εκατομμυρίων. Αλλά νομίζω ότι η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καλή. Δεν είμαστε στα πλαίσια συμβιβασμού. Εγώ θέλω να τοποθετηθώ σε αυτό το συμβαστικό πνεύμα και να σα προτείνω σαν εισηγήτρια να κρατήσετε μια γραμμή πιο φιλόδοξη, την πιο φιλόδοξη που γίνεται και μετά να υπάρχει και η βούληση συζητήσεις με το Συμβούλιο. Βέβαια, σε κάποια κράτη-μέλη, βέβαια, έγιναν προτάσεις με την ιδέα σταδιακής εφαρμογής phasing in με κατόφλιο που θα πρέπει να αποτελεί ένα σημείο ισορροπίας στη συζήτηση με το Συμβούλιο. Λαμβάνοντας υπόψη τις διεξαχθήσεις εργασίας του Κοινοβουλίου με το κείμενο από την Επιτροπή Πανά. Ε, νομίζω ότι ε, δεν πρέπει να επαναχωρήσουμε από τις θέσεις μας. Τώρα που χρειαζόμαστε ε, στεναρή θέση και εμπειρία που είχαμε, που ήθελε και το Κοινοβούλιο στο φυσικό τομέα, είναι μια προσέγγιση που δίνει αποτελέσματα. Κανεί δεν θα πει ότι διαβάζω όλα προσεκτικά τα κείμενα του Business Europe ε, όταν θέλουμε να συνεχίσουμε θέσει απασχόληση και επενδύσει στην Ευρώπη. Αλλά όταν ζητάμε δεν πρέπει να βγούμε τι προόδου στην, ε, στον τομέα. Έξοχη η έκθεση της Oxfam βάσει πληροφοριών επισήμων για τον τομέα. Αυτό χρησιμεύει σαν έλλειψη. Διότι στην έκθεση αυτή βλέπουν τραπεζικό τομέα δεν υπέφερε καθόλου πλευρά ανταγωνισμού όσον αφορά τι ε, απαιτήσει υποβολή αναφορών αναχώρα. Αντιθέτω, δόθηκαν εργαλεία η πρόοδος που επετέφθη πρόσφατα, πρέπει να πούμε, δεν θα είχε συμβεί άνευ των προσπαθειών της διαδικασίας BEPS ε του ΟΣΑ, αλλά άλλα θέματα, ανταλλαγή πληροφορία για τα φορολογικά, ελάχιστα πρότυπα και διαπίστωση ποιο είναι ο πραγματικό δικαιούχο ιδιοκτήτη. Όλα αυτά τα πρόθεσε όσα. Άρα είναι σημαντικό να μείνουμε όσο πιο κοντά μπορούμε στα πρότυπα αυτά του ΩΣΑ. το βαθμό του δυνατού να μην δυσχεραίνουμε το έργο του ΟΣΑ σε διεθνέ επίπεδο αν κινηθούν προ άλλη κατεύθυνση. Χρειάζεται σωστή ισορροπία. Τέλο, συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση συναδέλφων για τη ρήτρα διαφύλαξη. Είναι αναλογική, είναι ορθή, αν για, εμπορικά, για εμπορικούς λόγους θέλουν ε, να συζητήσουν με φορολογικέ αρχές και θέλουν εμπιστευτικέ πληροφορίε που δίνουν στι φορολογικέ αρχές για λόγους εμπορικούς, εμπορικής εμπιστευτικότητας, είμαστε ανοιχτοί και ευέλικτοι σε αυτό. Εξασφαλίζοντα όμως ότι για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ε, δημοσιοποιούνται ε, οι περισσότερες δυνατές πληροφορίε. Ευχαριστώ κ. Καλβέτη, έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε να μην καταγραστώ την καλοσύνη σας και να είμαι επικοδομητικό. Ε, όπως είπα πριν, ε, ξέρουν ότι το 10% των επιχειρήσεων είπαμε θα πάει στο 90% ε, αυτό θέλω να πει και ο συνάδελφος και να μην παραβλάψουν τα συμφέροντά μας με τις ρυθμίσεις. Μιλούμε τώρα για πληρωμή φόρου, άρα το πιο σημαντικό για τους επιχειρηματίες είναι ο όγκος, το ποσό του τζίρου με το οποίου θα καθοριστεί το πληρωτέο ποσό και γι' αυτό και είπαμε ότι 90% του τζίρου είναι ένα στοιχείο σημαντικό, δημόσιο. Για κάποιον που θέλει να ξέρει ότι η εταιρεία κινείται. Άρα αυτό το ποσό του τζίρου και δεν απαραίτητο να φτάσουμε και στις πιο μικρές επιχειρήσεις. Άρα πρώτα απ' το για την κυρία Μπερές, παρακαλώ να, να, να λάβετε υπόψη ότι αυτό που τα λέμε ε, το τα εννοούμε. Δηλαδή όταν θέλουμε συμβασμό, θέλουμε συμβασμό με την Επιτροπή. Αλλά όταν φτάσουμε στο 750 αυτό είναι απαράδεκτο λέμε. Ε, αυτό δεν είναι... Ε, συμβιβασμός. Θέλω συμβιβασμός γιατί θέλω να λάβει σάρκα και ωστά να μην καταπέσει αυτή η πρωτοβουλία. Γι' αυτό και συμφωνώ με την πρόταση της ε, του οπότε το 750 δεν με πειράζουν. Αλλά για να είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα, ας πούμε, πάμε στο 700, ε, στο 650 και ή συνάδελφοι που έχουν επιφυλάξει ε, ε, γι' αυτό λέω, γι' αυτούς λέω ότι χρειάζεται ένα συμβασμό. Ας πούμε, συνάδελφο Φεραγκό της Τάρας. Και λέμε ότι κοιτάμε προς τον ΩΣΑ για να φτάσουμε στο 90 τόσο του τζίρου. Ναι, θέλω συμβασμό. Αλλά εάν δεν είναι αυτό δυνατόν, εντάξει στις προτάσεις της Επιτροπής. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ζήτησα και εγώ το λόγο. Είναι περασμένη όμως η ώρα και θα περιοριστώ στις τοποθετήσεις μου ως εισηγήτρια. Ε, δουλεύουμε προς όλο ταχώς. Ε, έχουμε την επόμενη εβδομάδα και στο Στρασβούργο συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών και ο ΙΚΠΑΓΙΕ και οι υποφαινομένοι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συγκεράσουμε τις διαφορετικές θέσεις για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για το κατόφλι αλλά και για το περιεχόμενο των δηλώσεων. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθούμε παρατήρησα ότι όλοι προβάλλουν το ρόλο του ΩΣΑ και τον εξαιρετικό, την εξωτερική δουλειά που κάνει, το ξέρουμε πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, δουλειά μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να κάνουμε κάτι περισσότερο. Το reporting είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη διαφάνεια και με διαφύλαξη όρων ισότιμου ανταγωνισμού για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ακριβώς υποφέρουν από το γεγονός ότι οι μεγάλες κάνουν ό,τι θέλουν, γιατί δεν ξέρει κανείς από πού και προς τα πού μεταφέρονται, μεταβιβάζονται ποσά ε, έσοδα. Λοιπόν, σημειώνω πολύ σύντομα. Καλύτερη διαφάνεια. Δεν πρέπει να πλήττει τα συμφέροντα της επιχείρησης η διαφάνεια το είδαμε και με τις τράπεζες, ε, διαφάνεια, ε, δεν πρέπει να, πλή, να πλήξει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, κόστος ε, με μια εμφυή διαμόρφωσή του που να συνδυάζεται με τα κατάλληλα ε, στοιχεία, δημοσιοποίηση δηλαδή των απαραίτητων στοιχείων και κόστος των χαμηλότερο. Αυτά λοιπόν. Και τώρα ως Πρόεδρος επιτρέψτε μου να κήρυξω το πέρας της πρωινής συνεδρίας. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ όσους ε, έλαβαν το λόγο και έδειξαν διάθεση για συμβιβασμό εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ και ακόμη μια πολύ καλή σας μέρα.